Μια Ευρώπη βασισμένη σε αξίες και προσιλωμένη σε αποτελεσματικού δημοκρατικού θεσμού, η οποία προωθεί μια ευημερούσα οικονομία σε μια δίκαιη και συνεκτική κοινωνία. Ξεκινάμε αμέσως και να σας ενημερώσω ότι σύμφωνα με αυτήν την, κανόνα δεν έχουμε κάτι στη Ξεκινούμε. Πρώτη ομιλήτρια εκ μέρους των φιλελεύθερων, η Σοφία Ιντφέλτ για τέσσερα λεφτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συνάδελφοι. Πνέει άνεμος αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2016 και το 2017 θα καταγραφούν στα βιβλία της ιστορίας σαν χρόνια αναταραχής και ανανέωσης αναπροηγουμένου. Μεγάλη αύξηση των θρηστικών δυνάμεων χωρίς λύση. Βλέπουμε τα πρώτα σημάδια της Ευρωπαϊκής Άνοιξης όχι καλοκαίρι, μετά από χρόνια, από εντάσεις και δυσαρέσκεια, υπάρχει ένας, ε, ένας άνεμος προσδοκίας και αισιοδοξία. Όταν είχε συναντηθεί ο, ο κύριος ε, Μακρόν, τον κύριο Τρόμπ και τον κύριο Πούτιν, μιλούσε για μια Ευρώπη ε, Σουδέα. Σήμερα αισθανόμαστε ότι θέλαμε να προσχωρήσουμε και να εφαρμόσουμε και να είμαστε ηγέτε όσον αφορά την αλλαγή του κλίματο. Είμαστε περήφανοι για την Ευρώπη. Είναι αξίε που είναι κλειδί για την επανίδρυση τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Οι εκλογικέ εκστρατείε τα πρόσφατα χρόνια εστιάστηκαν όχι μόνο σε παραδοσιακά υλικά θέματα ασφάλεια ε, τη ε, θέσεων εργασία, κοινωνική ασφάλεια, αλλά πάνω σε αξίε πολιτισμού και ταυτότητα η παγκόσμια τάξη αλλάζει με μια ανευπροηγούμενη ταχύτητα και ο κόσμος ανησυχεί και έχει στεσαριστεί λόγω απώλειας ε, επικοινωνίας. Τα εθνικιστικά κόμματα έχουν ανταποκριθεί σπέρνοντα ε, το μίσο, την καχυποψία και το φόβο, υποσχόμενο ότι θα επιστρέψουν σε ένα φανταστικό παρελθόν. Εμεί αυτό το απορρίπτουμε. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η ανταπόκρισή μα στα σαφή ερωτήματα και τα θέματα τη αξία του πολιτισμού και τη ταυτότητα, οι απαντήσει που δώσαμε είναι επαρκή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια βαθιά πολιτική ένωση. Οι πρώτοι πολιτικοί έχουν κουραστεί προσπαθώντα να εξηγήσουν αυτό. Δεν θέλουν να το εξηγήσουν στου ψηφοφόρου. Παρουσιάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν τεχνοκρατική οντότητα που μπορεί να συνοψιστεί από πλευρά οικονομικών ωφελών ή κόστου. Αν ανησυχεί ο κόσμο για την απώλεια τη ταυτότητα, η κατάργηση των τελών περιαγωγή δεν θα του καθησυχάσει καθησυχάσει. Αν φοβούνται ότι απειλείται ο πολιτισμό του, η μείωση τη γραφειοκρατία δεν θα καθησυχάσει του φόβου του. Εάν είναι αβέβαιο ο κόσμο για τι κοινέ αξίε των κοινοτήτων μα, δεν θα βρουν κάποια άνεση σε εμπορικέ συμφωνίε και ανακούφιση. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε το πονοπόλιο καθορισμού των κοινών μα αξιών και τη ταυτότητά μα στου εθνικιστέ αυτό το καιρό τη μεγάλη αβεβαιότητας, της ανασφάλεια και τη αναταραχής στην κοινωνία δεν είναι εύκολο να υπερασπιστούμε τι κοινέ μα αξίε. Δεν έχουμε καθορίσει τι κοινέ μα αξίε ε, μόνο και μόνο για όταν οι εποχέ είναι καλέ, αλλά όταν είναι δύσκολοι οι καιροί, χαλεποί και όταν πρέπει να δοκιμαστούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο μια οικονομική δύναμη, αλλά έχει και μεγάλη ηθικό βάρο στον κόσμο. Μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι. Οι αξίε μα έχουν εμπνεύσει πάρα πολλού στον κόσμο και πολλοί άνθρωποι ονειρεύονται να ζούσουν σε μια ελεύθερη, δίκαιη και σταθερή και δημοκρατική κοινωνία όπω είναι η δική μα στην Ευρώπη. Τόσο πολύ που άλλοι βλέπουν τις αξίες μας σαν μια απειλή, κάτι που προσπαθούν να καταστρέψουν. Τα ελακιστικά κόμματα σε όλο τον κόσμο έχουν θεματολόγιο που βασίζεται σε εθνικισμό, ξενοφοβία, ομοφοβία και σεξισμό και κινούνται, και κινούνται κατά της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και του κοσμικού κράτους και πάνω απ' όλα απορρίπτουν τον πλουραλισμό και διατείνονται ότι υπάρχει ένας λαός, μία φωνή, μία αλήθεια και μόνο αλλά σαφώς οι πρόσφατες εκλογές έχουν αποδείξει ότι αυτό είναι σφαλμένο. Οι Ευρωπαίοι δεν θα μειωθούν σε μονοσδιάστατη καρικατούρα. Αν θέλουμε η Ευρώπη να γίνει ισχυρή, θα πρέπει να προωθήσουμε το αντίθετο. Θα πρέπει να προωθήσουμε την ποικιλομορφία, την Ευρωπαϊκή Ένταξη, Ένωση, την ισότητα και τον πλουραλισμό. Αυτό είναι το όλο ιστορικό, το υποβαθρό και νομίζω ότι το tweet του Μάνφρεντ Μπέμπερ που δεν είναι εδώ την περασμένη εβδομάδα δυστυχώ ήταν κάπω ε, παραπλανητικό, διότι έλεγε ότι ταυτότητα της Ευρώπης είναι πάνω απ' όλα χριστιανική. Όποιο το αρνείται αυτό, αρνείται την πραγματικότητα. Αλλά αγαπητέ συνάδελφοι, κύριε Βέμπερ, η πραγματικότητα ποια είναι. Η πραγματικότητα είναι ότι η πραγματική ψυχή τη Ευρώπη είναι η ποικιλομορφία τη και η ελευθερία τη επιλογή την να πιστέψει κανεί και ποιο είναι. Η δημοκρατία, το κράτο δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, ολοκληρώνω Πρόεδρε, δεν είναι απλώ ιδεώδη, αλλά είναι κεντρική σημασία για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση ω τομεί τη πολιτική. Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι προπόθεση για σταθερό κλίμα για επενδύσει και για ανάπτυξη. Ο σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων ζητική σημασία για την κοινή πολιτική μετανάστευση και την αστυνομική συνεργασία και το κράτο δικαίου είναι απόλυτα ουσιαστικό για την εσωτερική αγορά και την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Εν συντομία, οι αξίε είναι το κλειδί για μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ενώση και γι' αυτό η Άλντε βάζει πρώτη, τις πρώτες τις αξίες. Ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρους του Συμβουλίου η κυρία Υπουργό, η κυρία Ντάλη. Πρόεδρε, Επίτροπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δίνετε σήμερα να παρέμβω σε αυτό το επίκαιρο θέμα. Πρόκειται όντως για μια εποχή βαθύ, βαθέως στοχασμού για το μέλλον της Ευρώπης. Είναι χαρά μου λοιπόν που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να ακούσω τις απόψεις σας. Ο τίτλος αυτής της συζήτησης μας ε, δείχνει μια Ευρώπη που αρέσει σε όλους. Σε αυτήν οι αξίες έχουν κεντρική σημασία. Έχουμε δημοκρατικούς θεσμούς και έχουμε τον ειλικρινή στόχο να βελτιώσουμε τη ζωή και την ευημερία των πολιτών μας, όχι μόνο των λίγων και τυχερών, αλλά ολόκληρης της κοινωνίας. Αυτή η περιγραφή δεν απέχει τόσο πολύ από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε σήμερα και σίγουρα συνάδει με τις φιλοδοξίες που ξεκάθαρα έχει η Ευρώπη. Όμως παρόλα αυτά, μέχρι πριν από μερικούς μήνες οι προσπάθειες της Ευρώπης είχαν χάσει την αξία τους, είχαν απαξιωθεί και ε, τις αγνοούσαμε. Είτε διότι η Ευρώπη θεωρείται ότι έκανε πολύ λίγα ή ότι έκανε πάρα πολλά, παραπάνω από όσα έπρεπε. Πρόσφατα όμως φαίνεται ότι υπήρξε μια μεταστροφή στις αντιλήψεις για την Ευρώπη. Αντί να θεωρείται η Ευρώπη η πηγή όλων των δεινών, θεωρείται ένα μέρος της λύσης. Έχουμε κάποια θετικά μηνύματα ανανέωσης της εμπιστοσύνης και της υποστήριξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ίσως διότι ο κόσμος γύρω μας αλλάζει και οι εναλλακτικέ ε, σιγά σιγά χάνουν τη λάμψη τους. Ίσως έχουμε ξεκινήσει να συνειδητοποιούμε ότι η λαϊκιστική ρητορική υπεραπλουστεύει περίπλοκα ζητήματα. Και αυτό έχει αρχίσει να δείχνει τα ωριά του. Ίσως επίσης έχει αναγνωριστεί πλέον ότι η συνεργασία σε παγκόσμιες προκλήσεις όπως το εμπόριο, το κλίμα και η τρομοκρατία είναι καλύτερη από το να είναι κανείς μόνος του. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι όσο περισσότερο αισθανόμαστε πως είναι ότι απειλούνται οι αξίες μας, τόσο πιο πολύ θέλουμε να τις υπερασπιστούμε. Και με αυτόν τον τρόπο παίρνουμε μια νέα όθηση. Θέλουμε πιο πολύ, με μεγαλύτερη ορμή, να επιδιώξουμε τους στόχους μας. Ένα κοινό όραμα για ένα κοινό μέλλον εμπεριέχει ακριβώς αυτή την κοινή επιδίωξη στόχων. Στο μέλλον, λοιπόν, η Ευρώπη δεν θα πρέπει να επιβάλλει το όραμά της στους πολίτες. Αν δεν έχει την υποστήριξή τους, ε, δεν μπορεί να έχει επαναστατικές ε, ε, δράσεις και ιδέες. Ε, πρέπει η Ευρώπη να συμπεριλάβει τους πολίτες στις διαδικασίες της, να τους κάνει να αισθανθούν ότι ακούγεται η άποψή τους, ότι έχει νόημα αυτό που λένε. Και γι' αυτό με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε τη Λευκή Βίβλο η οποία θα εκινήσει μια ειλικρινή σκέψη και ε, διαδικασία σκέψης ε, και θα ξεκινήσει έναν ειλικρινή διάλογο. Επίσης, να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις συνεχείς προσπάθειές του να διασφαλίσει ότι ακούγονται οι απόψεις των πολιτών μαζί με την Κομισιόν θα έχετε κι εσείς με μερίδιο σε μια σειρά συζητήσεων για το μέλλον της Ευρώπης που θα γίνουν σύντομα. Εμείς στο Συμβούλιο ξεκινήσαμε μετά το Brexit να Μπαίνουμε και εμείς σε αυτή τη διαδικασία περισυλλογής στην Πρατισλάβα το Σεπτέμβριο σε άτυπη συνάντηση. Χαράξαμε ένα συγκεκριμένο οδικό χάρτη για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις πιο αδύρυτες ανησυχίες των πολιτών. Υπάρχουν ε, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την μετανάστευση, την τρομοκρατία, την οικονομική και κοινωνική ανασφάλεια. Καθώς ε, προχωρούμε σε αυτό το δρόμο, το Μάρτι, με την 60η επέτειο από τη συνθήκη της Ρώμης, είχαμε άλλη μια ευκαιρία να σκεφτούμε το κοινό μας μέλλον. Η ατζέντα που βγήκε από αυτό είναι ακριβώς η εγγύηση ότι θα επιδιώξουμε τους πιο σημαντικούς στόχους μας τα επόμενα δέκα χρόνια. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκτοτε έχει επικεντρώσει την ε, δουλειά του σε αυτές τις προτεραιότητες έτσι ώστε να έχουμε απτά αποτελέσματα και να πραγματώσουμε τις υποσχέσεις μας. Μέσα στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας της Λευκής Βίβλου, το Συμβούλιο λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα πακολουθητικά έγγραφα της Κομισιόν για να μπορέσει ε, να υπάρχει μια αξιόλογη συνεισφορά στη συζήτηση. Επίσης, ε, το έγγραφο για την παγκοσμιοποίηση δίνει ε, τις κατευθύνσεις για το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, στα θέματα παγκοσμιοποίησης και εμπορίου. Να σας πω συγκεκριμένα πράγματα. Η περισυλλογή για το μέλλον της Ευρώπης είναι μια μικροσκελής διαδικασία που απαιτεί χρόνο και την ανοικοδόμηση ε, εμπιστοσύνης. Δεν θέλουμε να ρισκάρουμε, να προσφέρουμε πρόωρα αποτελέσματα και τελικά να μην εκπληρώσουμε πλήρως τις προσδοκίες. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συνεχίσει να δίνει έμφαση στα απτά αποτελέσματα έτσι ώστε η προστιθέμενη αξία της Ευρώπης να φανεί και πρακτικά. Σε αυτό το πνεύμα η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης ε, θα δώσει μια νέα ορμή έτσι ώστε το Συμβούλιο να πραγματώσει βασικές ε, κεντρικές πολιτικές αντί να μείνει στη θεωρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα έχουμε τον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, τον κύριο Τίμερμαν. Ευχαριστώ. Θα χρησιμοποιήσω τα τρία λεφτά που μου δίδεται για να ε, προβληματιστώ για το έπαιξε η κυρία Ιντβέλτ στην εισαγωγή τη. Γιατί έθιξε το θέμα των θεμελιωδών αρχών με έναν τρόπο ε, πολύ σαφή και συνοπτικό. Ε, Επίση, απέρριψε τι λύσει ε, που προσφέρουν οι ακραίοι, οι εξτρεμιστέ, οι εθνικιστέ και οι ξενόφοβοι. Όμω, η ερώτηση παραμένει γιατί τόσοι πολλοί Ευρωπαίοι παραμένουν, ε, νιώθουν έλξη από αυτά τα ακραία και εθνικιστικά φαινόμενα ε, και κινήματα τα οποία έχουν και θα συνεχίσουν να έχουν ισχύ ε, εκλογικά εκτός και αν αντιμετωπίσουμε τις αιτίε. Πολλοί από τους πολίτες μας ανησυχούν γιατί φοβούν ότι χάνουν τη θέση τους. Είναι η πρώτη γενιά που φοβάται ότι τα παιδιά τους θα είναι σε χειρότερη θέση από τη ίδια. Φοβούνται εξαιτία των απειλών του τζιχαντιστικ, της τζιχαντιστικής τρομοκρατίας, γιατί έτσι σαν να χάνουν ταυτότητά τους και τις ελευθερίες τους. Φοβούνται διότι ε, στην παγκόσμια σκηνή ε, χάνεται η σταθερότητα και η ειρήνη. Ε, δείχνουν να χάνουν, ε, φοβούνται γιατί χάνουν την ισχύ τους. Συνεπώ δεν είναι μόνο η θεμελιώδεις αξίες αλλά και αυτοί οι φόβοι οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και μπορούμε να τι αντιμετωπίσουμε μόνο αν σταθούμε ενωμένοι ω Ευρωπαίοι. Ε, μαζί με τι αξίε μα, λοιπόν θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να προωθούμε ευρωπαϊκέ λύσει σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια προβλήματα. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στου πολιτέ μα ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν παραμείνουμε ενωμένοι. Αυτό είναι δύσκολο βέβαια. Μια εποχή που οι πολιτικές ε, ε, περί της ταυτότητας, οι ε, συζητήσεις της ταυτότητας ε, μονοπολούν την ατζέντα σε όλη την Ευρώπη. Δεν θα πρέπει να μιλούμε μόνο για την εσωτερική αγορά και το ενιονόμισμα, ε, ούτε μόνο για τη γραφειοκρατία. Αυτά είναι μέσα, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Σημαντικά μέσα, σημαντικά εργαλεία, αλλά έχουν νόημα μόνο αν βασίζονται στις κοινέ μας αξίες. Και δυστυχώς δεν μιλάμε αρκετά για αυτές τις αξίες μας. Το ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι οι άνθρωποι στους οποίους, στους οποίους επιτέθηκε η κυρία Εντβέλτ ε, εξαιτία του ότι δεν προσφέρουν λύσεις αλλά και δεδομένου ότι οι προτάσεις δεν είναι σοβαριστικής αξίας ε, αυτό, αυτό που έχουν όμως είναι ότι ξεκινούν από αξίες, ξεκινούν από ηθικά επιχειρήματα. Έτσι θα πρέπει να ξεκινήσουμε κι εμείς. Από τις αρχές οι οποίες έκαναν μεγάλη την Ευρώπη, κράτος δικαίου, δημοκρατία, πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό, αυτή είναι η τριπλέτα πάνω στην οποία έχει χτιστεί η Ευρωπαϊκή Συνεργασία. Και ο εξυγχρονισμός της στην μεταβιομηχανική εποχή σημαίνει ότι θα δημιουργηθεί μια κοινωνία πολυφωνική που θα δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες, περισσότερες φιλοδοξίες στους ανθρώπους, ε, θα διορθώσει την οικονομία στην μεταβιομηχανική περίοδο, ε, αλλά όλα αυτά θα γίνουν μόνο αν στηριχτούμε στις αξίες μας. Αυτή είναι και η βάση της Λευκής Βίβλου της Κομισιόν, όλων των αναλύσεων που έχουμε κάνει ως Κομισιόν και που θέσαμε στο τραπέζι ως κίνηση, σημείο κίνησης της συζήτησης με το Κοινοβούλιο αλλά και με τα κρατη ελπίζοντας ότι τα μέλη του Συμβουλίου θα χρησιμοποιήσουν αυτή τη βίβλο για να ξεκινήσουν και ένα διάλογο στο εσωτερικό τους, στα ίδια τα κράτη-μέλη. Τελειώνοντας, να πω το εξής. παρατηρούμε ότι ξυπνά μια καινούργια γενιά στην Ευρώπη με τις Βρετανικές ε, εκλογές, με τις Γαλλικές εκλογές, με τις πορείες των γυναικών στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Γιατί? Γιατί τώρα καταλαβαίνουμε πως ε, παρόλο ότι οι αξίες μας είναι σαφείς ε, και είναι, ε, είναι και αιώνιες και δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, δεν μπορούν να καταστραφούν. Αλλά παρόλο ότι είναι σαφείς και παρόλο ότι είναι η βάση της συνεργασίας μας, αυτές οι αξίες, βλέπουμε σε όλο τον κόσμο ότι αυτές οι αξίες δεν είναι ε, ε, ε άθραυστες χρειάζεται να τις προσπίσουμε. Και εδώ δεν είναι θέμα αριστεράς ή δεξιά. Είναι το θέμα αν επιλέγουμε μια ανοιχτή κοινωνία όπου όλοι συμμετέχουν και κανένα δεν μένει εκτό, ή θα, πέσει, θα πέσουμε στην παγίδα του να πιστεύουμε ότι τα αδέλφια μα είναι και εχθροί μα. Εμεί θέλουμε μια ανοιχτή κοινωνία που όλοι έχουν την ίδια αξία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Αντιπρόεδρο. Και τώρα ερχόμαστε στον κατάλογο των ομιλητών. Για 1,5 λεπτό η Ρόζα Εστάρα Φέραγκουτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν από 60 περίπου χρόνια, στις 25 Μαρτίου ε, του 1957, οι Ευρωπαίοι υπέγραψαν την ε, συνθήκη της Ρώμης ε, και έσπηραν το σπόρο της Ευρώπης. Ε, κάτι που οδήγησε σε μια μεγάλη περίοδο ευημερίας και σταθερότητας και ε, ελευθερίας. Ο Σούμαν τότε είχε πει ότι η Ευρώπη δεν θα γίνει διαμιάς, ε, αλλά σιγά σιγά, σταδιακά, με μικρά επιτεύγματα που θα καλλιεργούσαν την αξία της ελεγγύης. Τότε, εκείνη την εποχή, η πατέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν, ε, δεν είχαν σαφή το στόχο της Ενωμένης Ευρώπης, αλλά μας, ε, απέδει, μας ε, έδειχναν ποιοι είναι οι εχθροί. Ε, ο εθνικισμός, η γενοκτονία, ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, η πόλεμη και ο ολοκληρωτισμός. Σήμερα η Ευρώπη έχει αλλάξει, έχει ενηλικιωθεί. Ε, ε είμαστε λιγότεροι εμείς αλλά δεχόμαστε περισσότερη μετανάστευση. Έχουμε το πρόβλημα της ανεργίας. Έχουμε προκλήσεις όπως η μετανάστευση, η ασφάλεια, η ενέργεια, η οικονομία, η άμυνα. Ε, είναι μια περίπλοκη Ευρώπη, ε, γεμάτη αντιθέσεις. Έχουμε την, την πρόκληση της πολυφωνίας και της ένταξης όπως είπε ο Επίτροπος, ε, η πρόκληση όμως, η πραγματική πρόκληση είναι να μείνουμε ενωμένοι. Η ελευθερία, ε, η, η, ειρήνη και η πρόοδο θα πρέπει να παραμείνουν στόχοι, αλλά αυτό θα πρέπει να το, πιστέψουμε. Και αυτό όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στην πράξη. Ευχαριστώ. Τώρα για δύο λεπτά η κυρία Τάνια Φαγιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο τίτλος σημερινής μας συζήτησης είναι η επανίδρυση, αν της Ευρώπης. Έχουμε πλήρη επίγνωση ότι τα θεμέλια καταραίουν και ότι η δημοκρατία, η ισότητα και ο σεβασμός είναι αυτά τα θεμέλια. Και ο σεβασμός, κύριε Αντιπρόεδρε Τίμερμαν, αναφερθήκατε σε αυτό στη ρητορική των λαϊκιστών και την οργή των πολιτών μας. Τα πνευματικά λοιπόν η λύθη, η πνε, πνευματικοί καταραίων του οικοδομήματος. Και αυτό το βλέπουμε όταν δεν λαμβάνουμε υπόψη και δεν εφαρμόζουμε τι προσωστώσει των προσφύγων. Λαμβάνονται αποφάσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω, αλλά δεν εφαρμόζονται από κάποια κράτη-μέλη. Γι' αυτό καλωσορίζω την απόφαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει η διαδικασία επιπαραβάση κατά των κρατών μελών εκείνων που δεν συμμετέχουν ε, στον επιμερισμό του άχθου. Χθε συζητήσαμε εκθέσει για τη Σερβία και το Κωσυφοπαίδιο, που περιμένουν στην αίθουσα αναμονή για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε πάρα πολύ αυστηροί όταν θέλουμε να παρακολουθούμε και να κρίνουμε την εφαρμογή των κριτηρίων τη Κοπενχάγη. Αν αυτέ οι χώρε δεν πληρούν τα κριτήρια, ποτέ δεν θα γίνουν κράτη-μέλη. Πιθανότατα αυτή είναι και μια δίκαιη τιμωρία. Είναι όμω σωστό και δίκαιο η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει αυτή την κρίση που έχει κάποια κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που ε, δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια. Ποια είναι η τιμωρία αυτές τι χώρες που συμμορφώνονται με αυτά τα κριτήρια. Αυτό λοιπόν χρειάζεται δημοκρατία και αλληλεγγύη να εφαρμόζεται παντού και ελευθερία. Και πρέπει να επικρατεί δικαιοσύνη. Ε, προκαιρού στους σοσιαλιστές S&D υποστηρίξαμε την ιδέα της δημιουργίας ενός συστήματος βαθμολόγησης δημοκρατίας με δείκτες αξιών. Εγώ συμφώνησα με αυτή την πρόταση. Ε, ταυτόχρονα όλοι γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση. Ώρα έχουν μετρηθεί, τίποτα όμως δεν θα αλλάξει όσο οι παραβάτες δεν τιμωρούνται. Δεν αληθεύει το ότι δεν έχουμε μηχανισμούς. Δεν θέλουμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Για ένα λεπτό, Ρόμπερτ Τσίλε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν ήθελα να διαβάσω το τίτλο, αν διάβασα τον τίτλο, είναι τόσο μακροσκελή, θα τελείωνε ο χρόνο αγόρευση. Όταν βλέπουν τέτοιου τίτλου και ονομασίε οι πολίτε, δεν μπορούν να καταλάβουν και απλησιάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που θέλουν οι διαοί μα θέλουν να δουν κάτι εύληπτο, να καταλάβουν πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτω ώστε οι αξίες που όλοι υποστηρίζουμε και όλοι αναφέρουμε να μην είναι κάτι ε, δυσνόητο για αυτούς και να μην είναι κάτι αντίθετο με τις αξίες των χωρών τους. Αν κάθε φορά χρειάζεται, δίνουμε διαφορετικές ερμηνείες και δίνουμε πληροφορίες που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, αυτό δεν βοηθάει. Γι' αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο συζητούμε και παρουσιάζουμε τα θέματα αυτά. Θα πρέπει να μπούμε σε μεγαλύτερο βάθος για να υπάρχει καλύτερη κατανόηση. Αν θέλουμε να μιλήσουμε κοινωνική συνοχή, ο κόσμος θέλει να είναι ανταγωνιστικός, αλλά και θα πρέπει να προσέχουμε να έχουν σωστή προσέγγιση και παρουσίαση των θεμάτων. Ευχαριστούμε. Για ένα λεπτό ο κύριος Παγκάτσαρ Η κυρία. Εγώ είμαι ε, ελάχιστα αισιόδοξη όπως και η κυρία Ιντβέλτ γιατί οι εθνικιστές και οι λαϊκιστές ε, δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι μια καινοτομία έχουμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε ε, την αχίλιο πτέρνα τους ε, ε σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία βέβαια υπάρχουν, υπάρχει τόση ομίχλη που πολλές ε, φορές ο ευρωπαϊκός ε, φάρος ε, δεν είναι ορατός. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να κάνουμε αυτό που είπατε εσείς καταρχήν, αρχές, θεμελιώδεις αρχές. Και για αυτές θα πρέπει να είμαστε ακέραιοι και ε, θαραλέοι. Μόνο και επίσης θα πρέπει αυτά που λέμε να συμπίπτουν αυτά που κάνουμε. Με άλλα λόγια δεν μπορούμε ε, να εντάξουμε στην Ευρώπη όλους αυτούς τους νέους που ε, θέλουν μέλλον, θέλουν ευκαιρίες και τους οποίους έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια. Τους χρειαζόμαστε, χρειαζόμαστε κυρίως τους νέους. Χρειάζεται να τους δώσουμε θέσεις εργασία και δικαιώματα. Θα πρέπει και αυτοί να είναι το ίδιο παθιασμένοι με εμά για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Thank you Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος, επόμενος, επόμενη ομιλήτρια για ένα λεπτό, Ματίνα Άντερσον. Το Brexit, Brexit ήταν αφύπνιση. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια κοινωνική Ευρώπη που θα βασίζεται στη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και μια εθνική προοδευτική κυριαρχία. Αντί όμως να ακούμε όλα αυτά, ακούμε ε, πολλά για μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων, αλητότητα, έναν ευρωπαϊκό ε, στρατό. Νομίζω ότι είναι λάθος. Ε. Το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι περισσότερη ενωμένη Ευρώπη με περισσότερα κονδύλια προς αυτές τις κατευθύνσεις. Ο κόσμος θέλει περισσότερη αλληλεγγύη και περισσότερη δημοκρατία, όχι διάσωση των εταιριών. Δεν πρέπει να αγνοούμε αυτές τις επιταγές για δημοκρατία γιατί πρέπει να προστατεύσουμε ε, όλες τις ε, συμφωνίες βάσει των ΗΕ, Το Sinn Féin πιστεύει σε μια Ευρώπη που θα αντιμετωπίζει ισότιμα όλα τα μέλη, όλα τα παιδιά. Κανείς δεν θα αγνοείται και πραγματικά ε, πολλοί από εμάς εδώ δεν έχουν κατανοήσει αυτό το στόχο. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα για ένα λεπτό, Raymond Finch. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, μιλήσατε για την επαναθεμελίωση της Ευρώπης βάσει αξιών που έχουν να κάνουν με αποτελεσματικούς ε, δημοκρατικούς θεσμούς ε, που υποστηρίζουν μια ευημερούσα κοινωνία. Εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζουμε το ταξίδι μας προς την ανεξαρτησία. Η θεώρηση της Ευρώπης που έχουμε εμείς είναι τελείως διαφορετική. Βασίζεται στην, ε, στις ευκαιρίες, στον νεοαπικιοκρατισμό και σε ε, θεσμούς που είναι τελείως αντιδημοκρατικοί. Οδηγούν στην ανέχεια, το διχασμό και πραγματικά σε καταστροφή ε, στον νότο της Ευρώπης και στις οικονομίες του. Θεωρείτε ότι αυτή η καταστροφή όπως το 40% των νέων ανέργων στην Ευρώπη θα μπορέσει να αντισταθμιστεί με το Eurorail. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο, πολύ κακό να βάζουμε γύψο σε μία ανοιχτή πληγή. Ο μόνος τρόπος που μπορούμε να επιτύχουμε την σταθεροποίηση είναι να ακολουθήσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα, ε, Άλκη Ζέστρα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, οι ευρωπαϊκές αξίες πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που τα κράτη-μέλη και ε, οι πολίτε των κρατών μελών έχουν διαφορετική άποψη από τις Βρυξέλλε. Θα πρέπει λοιπόν να είναι σωστή προσέγγιση όσον αφορά την ασφάλεια και τη μετανάστευση και άλλα θέματα θα πρέπει να έχουμε τα κατάλληλα μέσα να καταπολεμήσουμε το λαϊκισμό και να αντιμετωπίσουμε την όλη κατάσταση που δημιουργείται. Υπάρχει και το θέμα τη ε, Τουρκία, η κατάσταση στην Τουρκία και έχουμε και το Ηνωμένο Βασίλειο που θέλει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Χρειαζόμαστε μια νέα βάση συνεργασία, ευρωπαϊκή συνεργασία, μια συνεργασία η οποία ίσω να στεφθεί από επιτυχία αν τα κράτη-μέλη ε, ξαναβρούν το κύρο του, ε, όταν τα εθνικά κοινοβούλια εκ νέου ε, το σωστό του ρόλο. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εξαφανιζόταν σε αυτή την περίπτωση. Θα, έτσι θα κάναμε μισό δισεκατομμύριο ε, σε έξοδα. Τώρα για ένα λεπτό ελευθέρω συναδεινός. Είναι πλέον απαραίτητη η σύγκληση συνεδρίου αναμόρφωσης και επανεθεμελίωση με εντολή τη μεταρρύθμιση τη Ένωση και το κοινό μέλλον εθελοντικά συνεργαζόμενων κυρίαρχων κρατών με στόχο την ανακατανομή και επαναπατρισμό αρμοδιοτήτων Έω τότε ο τρόπο λήψη αποφάσεων στο ευρωπαϊκό συμβούλιο εάν δεν προβλέπεται ομοφωνία πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά στη βάση τη διπλή ενισχυμένη πλειοψηφία ω προ τον αριθμό κρατών μελών και του συνολικού πληθυσμού τη Ένωση. επιπλέον όσον αφορά στην επιτροπή πρέπει να αντιμετωπιστεί το εγγενές δημοκρατικό έλλειμμα υπό την ισχύουσα διαδικασία τη κομιτολογία δια τη συμμετοχή των αρμοδίων υπουργών και τη δημοσιοποίηση των θέσεων και των ψήφων του. η μελλοντική ένωση πρέπει να είναι λειτουργική βιώσιμη και δημοκρατικά αποδεκτή και όχι ένα ξέπλυμα του σημερινού αναποτελεσματικού και διαφανούς μοντέλου. με διακυβερνητικέ διαδικασίε και λαμβάνοντα υπόψη τι εθνικέ ανάγκε των κρατών μελών να επικεντρωθεί σε ζητήματα με πραγματικά διευρωπαϊκό διασυνοριακό πρόσημο όπω η κλιματική αλλαγή ή η αποτροπή μετακίνηση εκατομμυρίων λαθρομεταναστών από την υποσαχάρια αφρική και την ασία προ την ευρώπη. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα για 1,5 λεπτό Κάρλος Κουέλιο. Ο Πούτιν επέστρεψε στον ψυχρό πόλεμο ε, και δηλητηριάζει την κοινή μας νόμη, ε, ε, στρατιωτικοποιεί τα σύνορα. Ε, οι λαϊκισμοί κερδίζουν έδαφος, αλλά τελικά χάνει το, τις εκλογές από την Ολλανδία μέχρι την Αυστρία, στην Γαλλία, ακόμα και στις τελευταίες Βρετανικές εκλογές. Γιατί, όπως έλεγε ο Ρόμπερ Σούμαν, η Ευρώπη κάνει συγκεκριμένα βήματα, συγκεκριμένα επιτεύγματα και η δική μας Ευρώπη είναι κάτι παραπάνω από ένα οικονομικό κατασκεύασμα. Είναι ένα όραμα κοινή ηθαγένειας. Ε, μια ολόκληρη γενιά έχει μεγαλώσει. Η Ευρώπη είναι, με αυτόν τον τρόπο η Ευρώπη είναι η Συμφωνία του Παρισιού, η Ευρώπη είναι ο ουμανισμός, η Ευρώπη είναι Σέγγεν, η Ευρώπη είναι η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων που κινούνται ελεύθερα μέσα σε, μια, σε ένα ωκεανό ευκαιριών. Η Ευρώπη είναι το πρόγραμμα 2020. Ε, είναι η Ευρώπη της τεχνολογίας που σώνει ζωές. Αυτή είναι η Ευρώπη στην οποία πιστεύω. Η Ευρώπη των ανθρώπων, η Ευρώπη των πολιτών. Και δεν χρειάζεται ε, να ε, ξαναστηθεί η Ευρώπη ε, σε καινούριε βάσεις. Η Ευρώπη έχει βάσεις. Η Ευρώπη είναι οι δικές μας δεσμεύσεις με η προσήλωση στην ελευθερία, στα δικαιώματα, στην ευημερία. Θα πρέπει να επαναβεβαιώσουμε την πίστη μας στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κοέλιο. Και τώρα για ένα λεπτό ο κύριος Νίντερ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Στην Ευρώπη υπάρχουν πάρα πολλές διαφωνίες ε, με τις οποίες είμαστε αντιμέτωποι. Έχει να κάνει με το μέλλον όλων μας. Ε, είμαστε σε ένα σημείο καμπής. Ήρθε η στιγμή λοιπόν να προχωρήσουμε πέρα από τον βιομηχανικό καπιταλισμό. Ε, υπάρχει ε, μια, ένας κοινωνικός κατακαιρματισμός, ε, η πολυπολιτισμικότητα, όλα αυτά τα στοιχεία που μας πάνε στον καινούριο κόσμο, στον οποίο δεν μας βοηθούν τα προηγούμενα γνωστά σενάρια. Πρέπει να φτιάξουμε μια νέα Ευρώπη, μια νέα Ευρώπη η οποία θα βασίζεται στην πρόοδο, την αλληλεγγύη, την ελευθερία και την ασφάλεια. Νομίζω ότι πρέπει να διαμορφώσουμε μια τέτοια Ευρώπη ώστε να μην ε, υφίσταται σε αυτή ο στιγματισμός ε, και το μίσος. Θέλουμε μια Ευρώπη όπου όλοι θα αισθάνονται σαν στο σπίτι τους, όπου δεν θα υπάρχει φόβος, αλλά μόνο ελπίδα και ευκαιρίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Νίτερ Μιούλερ και τώρα για ένα λεπτό σε Τσανέσκι. Κύριε Πρόεδρε, είμαστε πολιτικοί. Πρέπει να μιλάμε ειλικρινά ποιες ήταν οι επιτυχίες, η βάση της επιτυχίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα. Το ότι έξι χώρες και μετά αργότερα 10, 12, 15 χώρες εργαστήκανε βάση συνένεσης. Υπήρξε ένα ελάχιστο στο οποίο συμφωνούσαν και συνεργαζόταν οι χώρες σε ένα πνεύμα αλληλεγγύης. Κανείς δεν υποχρέωνε τίποτα, δεν πίεζε τον άλλον Γαλλία εναντίον των άλλων πέντε χωρών Φερρυπίν. Στην αρχή είχαν γίνει τις συζητήσεις. Υπήρχαν προβλήματα στην αρχή με την αγροτική πολιτική και αποφάσισαν να ακολουθήσουν μια κοινή πολιτική. Και είχαν αποφασίσει ότι δεν πρέπει να πλήττονται τα συμφέροντα καμιά χώρα για να προχωρήσουν. Πιστεύω λοιπόν ότι η βάση για την επιτυχία του ευρωπαϊκού εγχειρήματο είναι όταν δρούμε σε πνεύμα αλληλεγγύη, να υπάρχει συνένεση να μην ε, ψηφίζουμε και να καταπιέζουμε άλλες χώρες. Αλλιώς δεν θα λειτουργήσει. Ε, δεν υπάρχουν μπλε κάρτες. Σύμφωνα με τον κανόνα ε, με τον οποίο εργαζόμαστε, αυτό είναι ξεκάθαρο. Και τώρα Σίση Λιβίξτρομ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Σύμφωνα με το, Ευρωβαρόμετρο, οι πολίτες μας στηρίζουν την ευρωπαϊκή συνεργασία σε πολύ μεγάλο ποσοστό και όλο και περισσότεροι θέλουν μια πιο ε, ευρεία και πιο βαθιά συνεργασία στο μέλλον. Οι πολίτες μας πιστεύουν στο μέλλον της Ευρώπης και προφανώς αυτό θα πρέπει να μας εμπνέει στο, στην καθημερινή μας δουλειά. Ε, πολλά εκλογικά αποτελέσματα μεταξύ αυτών του Μακρόν στην ε, Γαλλία υποδεικνύουν την ανάγκη να ακολουθήσουμε μια κεντρώα πολιτική και θα πρέπει να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε την Ευρώπη. Πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Θα πρέπει να βρούμε λύσεις ε, σε διασυνοριακά προβλήματα που να κοιτούν στο μέλλον. Η ίδια δημοσκόπηση του Ευρωβαρομέτρου μιλάει ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε κοινέ λύσεις για την μετανάστευση, την τρομοκρατία και το κλίμα. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το μέλλον των πολιτών μα όλοι μαζί. Ευχαριστούμε. Και τώρα θα ακούσουμε για ένα λεπτό τον Κώστα Χρυσόγονο. Η ιδρυτική συνθήκη προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων ενώ διακηρυγμένος σκοπός της είναι να προάγει την ειρήνη και την ευημερία των λαών της. στην πραγματικότητα όμως η ένωση ανέχεται την παραβίαση των αρχών του κράτους δικαίου στην ουγγαρία και την πολωνία. παράλληλα η πολιτική λιτότητα που έχουν επιβάλει οι ισχυροί της ευρωζώνης οδηγεί σε συρρήκνωση θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων όπως τα δικαιώματα στην υγεία την κοινωνική ασφάλιση τη συλλογική διαπραγμάτευση τις δίκαιε συνθήκε εργασίας και τη δημιουργία οικογένεια, ιδίω στις χώρες του νότου όπως η ελλάδα. αν θέλουμε να αποκτήσει το εγχείρημα τη Ευρωπαϊκή ενοποίησης μακροπρόθεσμη προοπτική πρέπει να αποδείξουμε στην πράξη τον σεβασμό μας στις αξίες και τους σκοπούς της ένωσης και πρέπει να τον αποδείξουμε τώρα αλλάζοντα πολιτικέ πριν να είναι πολύ αργά. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα για δύο λεπτά, Πίτερ Λούντκρεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρώπη βασίζεται σε αξίες. Αυτό είναι το θέμα που συζητούμε σήμερα η ευθύνη μας ε, για τα χρήματα που δαπανούν ε, οι φορολογούμενοι είναι ακριβώς ο θεμέλιος λήθος ε, αυτής της συζήτησης για την επαναθεμελίωση της Ευρώπης. Ας πούμε, στο Βρυξέλλες έχουμε ένα κτίριο το οποίο τελείωσε το 1993 και κόστισε πάρα πολλά χρήματα. Αυτή τη στιγμή ε, πρέπει να το ξαναφτιάξουμε γιατί ε, ήδη έχει ανακαινιστεί πάρα πολλές φορές. Ε, το 2014 ήταν η τελευταία φορά. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν στο μέλλον να έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που να μοιάζει περισσότερο με το Αμερικάνικο Κογκρέσο. Δεν ξέρω αν αυτό αποτελεί μια, καλή, ένα καλό όραμα για ένα Ευρωπαϊκό σύστημα Ηνωμένων Πολιτειών ε, να έχουμε τόσο, τόσο ψηλό κόστος ε, πραγματικά ε, μας κάνει πολλές φορές να πανικοβαλόμαστε διότι τελικά τέτοιες αποφάσεις μπορεί πολλές φορές να οδηγήσουν τρεις φορές στο μεγαλύτερο κόστος. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα σωστά. Ε, το να χτίσουμε άλλο ένα τέτοιο κτίριο στι Βρυξέλλες νομίζω δεν είναι ο σωστό τρόπος. Πρέπει να έχουμε ακριβώ έλεγχο των, του τρόπου που χρησιμοποιούμε τα χρήματα των φορολογούμενών μας. Αλλιώς ε, ε, πραγματικά το να καταδαφίσει ένα ήριο 25 ετών είναι τρέλα, όπως και να το ανακαινίζεις. Ε, όλα αυτά ε, πραγματικά δεν ακούγονται ωραία στους Ευρωπαίους. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Λούντκριν. Και τώρα ένα λεπτό Γκέρκ Μάιερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι ευρωπαϊκές αξίες, ε, όπως υπόθηκε ήδη, στην ουσία ε, πώς ορίζονται, ποιος τις ορίζει εμείς. Νομίζετε ότι μπορούμε να το κάνουμε εδώ στην Ευρώπη. Οι άνθρωποι ούτε οι ίδιοι δεν μπορούν να τις ορίσουν. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές σε όλη την Ευρώπη. Αξιότιμοι συνάδελφοι, υπάρχει ποικιλομορφία. Αυτή την εκτιμούμε. Αλλά πολλές φορές τη φοβόμαστε κιόλα. Τα αποτελεσματικά δημοκρατικά θεσμικά όργανα είναι κάτι που όλοι υπογραμμίζουμε. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να έχουμε και αποτελεσματική αντιπολίτευση, όπως είπε και η κυρία Φαντ Συνήθω ε, ε, συνήθως ε, αυτή η αντιπολίτευση δεν υπάρχει. Πολλές φορές έχω την εντύπωση οι συνάδελφοι ότι όλοι από όλες τις πλευρές λέμε το ίδιο πράγμα και για τα ίδια πράγματα διαφωνούμε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα για ένα λεπτό Ζολταν Μπάλτσο. Ευχαριστώ. Η κυρία Ινφελτ μίλησε για κόμματα και τα χαρακτήρισε ως εθνικιστικά και ε, ε, έχει τη δική της προσωπική αλήθεια. Όμως ε, δεν είναι αυτή η οποία οποία ε, εκπροσωπεί τη μία και μοναδική αλήθεια. Όλοι αυτοί δηλαδή που είναι υπέρ της Ένωσης δεν είναι οι μοναδικοί που έχουν την αλήθεια και όλοι οι άλλοι πρέπει να καούν στην πυρά επειδή είναι αντιευρωπαίοι. Εμείς συζητούμε τις αξίες και ο Μάνφρετ Βέμπερ μίλησε για τις χριστιανικές μας ρίζες. Χρειαζόμαστε όμως και την ποικιλομορφία, την πολυπολιτισμικότητα Αυτά είναι μεταξύ των βασικών μας ε, θεμελιωδών μας αξιών, όπως είπε και ο Σούμαν. Η Ευρώπη ε, δεν ε, μπορεί να γίνει πιο ενωμένη παρά μόνο αν είναι ένας ο στόχος της και όσο πιο χριστιανική γίνεται τόσο πιο ενωμένη θα είναι. Αυτό το είπε ένας από τους πατέρες της Ευρώπης. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Ευχαριστούμε. Και τώρα για 1,5 λεπτό Τσάμπερ Σόγκορ. Κοιτάξτε, δεν πιστεύω εγώ ότι πρέπει να επανοικοδομήσουμε βάθρων την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χρειαζόμαστε μια επανάσταση πολλά από τα κακά που αποδίδουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πρώτη κάτι για το οποίο φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά γίνονται και προβολέ. Όπω είναι το θέμα του δημοκρατικού ελλείμματο. Μπορώ να πω σίγουρα ότι η νομοθετική διαδικασία τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω είναι πολύ πιο διαφανή, ελεγχόμενη και συμπεριλαμβάνει πολύ περισσότερου από αυτή που χρησιμοποιείται στη χώρα μου. Τούτου λεχθέντο υπάρχει περιθώριο για πιο ε, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αντοχή και καλύτερη ανταπόκριση προσδοκίες των πολιτών. Ήδη οι συνθήκε ε, που υπάρχουν τώρα προσφέρουν τι περισσότερε απαντήσει σε αυτά τα θέματα. Αυτέ οι απαντήσει όμω αγνοούνται πολύ συχνά. Βλέποντα το, το μέγεθο του τίτλου, και δεν θα μπορούσε να πει κανεί η συζήτησή μα δεν είναι φιλόδοξη θα πρέπει να επιμείνω επί των αξιών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 των συνθήκων. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποτίθεται ότι εδράζεται μεταξύ άλλων επί της αξίας της ισότητας, της μη διάκρισης και του σεβασμού της ποικιλομορφίας. Ακόμα έχουμε πολύ δρόμο να ακολουθήσουμε για να έχουμε αποτελεσματική προστασία αυτών των αξιών στο συγκεκριμένο τρομέα των ε, γλωσσικών μηνοτήτων ή των αυτοχθόνων, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αποφύγει τις διακρίσεις που έχουν αρνητικές συνέπειες όσον αφορά τη γλώσσα και τον πολιτισμό ανθρώπων που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες και τελικά ε, ε, βλάπτεται και η κυλομορφία της Ευρωπαϊκής Ενώσεω. Πάνω από 60 εκατομμύρια πολίτε περιμένουν την αποδοχή της ύπαρξής τους από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Σας ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σόγκορ και τώρα για ένα λεπτό Γιώ Λάινεν. E η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι περισσότερο από μια μεγάλη αγορά. Είναι μια πολιτική κοινότητα. Για πολλά χρόνια μαχόμασταν για αυτές τις αξίες. Το πολιτικό προφίλ της Ευρώπης πρέπει να γίνει πιο ορατό και να γίνει και πιο προοδευτικό. Αυτό το που είπε ο Αντιπρόεδρος είναι σωστό. Αυτές είναι οι αξίες για τις οποίες μαχόμαστε και όταν καταστρατηγείται η δημοκρατία ή η, η ελεύθερη έκφραση της άποψης του καθενός ε, δεν είναι σωστό. Οι πολίτες ε, πραγματικά ε, είναι αντιμέτωποι με περιπτώσεις όπου τα μισά κράτη-μέλη κάνουν τη ε, ε, δουλειά τους και τα άλλα απλώς παρατηρούν. Φαίνεται ότι είναι αδύναμα. Υπάρχει το dumping ε, στη φορολογία, αθέμητος ανταγωνισμός, εγκληματικότητα, πολλές πολιτικές που επιδεινώνονται. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα πέντε σενάρια στη Λευκή Βίβλο που θα οδηγήσουν σε ένα ενιαίο πρόγραμμα για τα επόμενα στάδια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Θα είναι από κοινού αυτή η προσπάθεια. η τρύπα για ένα λεπτό τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η επαναθεμελίωση μιας Ευρώπης που βασίζεται σε αξίες και σε δημοκρατικούς θεσμούς με μια ευημερούσα κοινωνία και οικονομία. Όταν διαβάζω αυτό τον τίτλο ε, σκέφτομαι τον χορό των ξωτικών ε, που ε, από μόνο τους χορεύουν και τραγουδούν. Νομίζω λοιπόν ότι το να φτάσουμε σε μια τέτοια ρίση είναι σαν να ομολογούμε την ε, αποτυχία μας. Είμαστε ε, στα όρια της κοινωνίας για με το θέμα του ευρώ, της μετανάστευσης, την πολυπολιτισμική κοινωνία. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λοιπόν, ε, δεν είναι ο κανόνας, δεν είναι η εξαρεσία, αλλά ο κανόνας τα προβλήματα. Πολλοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητούν ε, μια Ευρώπη ε, η οποία θα είναι όλο και πιο ενωμένη, πιο κεντρική, θα υπάρχουν κοινά σχέδια, περισσότερη γραφειοκρατία και πατερναλισμός. Ε, η απάντηση είναι λιγότερη απόδοση, λιγότερες παραδόσεις, λιγότερη πολυπολιτισμικότητα, λιγότερη δημιουργικότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Τρεμπέσιους και τώρα για ένα λεπτό Μαρίνα Άλμπιους Άλμπιους-Ούσμαν. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε αρχέ νεοφιλελεύθερης με τον έλεγχο του ελλείμματος, φιλελευθερωπιστών υπηρεσιών, ε, με αντιδημοκρατικά όργανα και ε, οικοδομημένη πάνω σε ένα σαφή στόχο, την κοινή αγορά. Αυτό δεν αλλάζει με κάποιε μικρομεταρρυθμίσεις, με μια λευκή βίβλο πολύ δε περισσότερο με αυτά τα που μας οδήγησαν στην ε, αύξηση της ακροδεξιάς, στο Brexit ε, ή στην αύξηση των ανισοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση του Ευρώ, ε, του, του Μάστριχτ, της αντιμετανάστευσης δεν μπορεί να αλλάξει με αυτόν τον τρόπο. Αυτό από την άλλη μεριά δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να οδηγηθούμε σε ρήξη με την Ευρώπη. Το αντίθετο. Εσείς θέλετε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση των ε, πολυεθνικών. Εμείς θέλουμε μια Ευρώπη για τα λαϊκά στρώματα. Με τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Πορτογαλίας. Όλοι μαζί και όλες μαζί. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό η κυρία Φων Στόρτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση σήμερα μιλά για την απενεθελημελίωση της Ευρώπης που βασίζεται σε αξίες και μια κοινά δομημένη κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι κάτι έχει καταρρεύσει για να το επαναθεμελιώσουμε και ε, ο κύριος Τίμερμανς μίλησε για τις αξίες της Ευρώπης, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Κανείς εδώ μέσα δεν είναι κατά αυτών των δύο ε, ε, αξιών. Όμως το πρόβλημα είναι και τώρα γελάτε επειδή ε, κανείς υπερασπίζεται την εθνική κυριαρχία θεωρείται ότι δεν είναι δημοκράτης και ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Αυτό είναι παράλογο και φέρνει τις χώρες αντιμέτωπες τη μία με την άλλη. Θέλουμε αξίες. Σας θυμίζω ε, τον ε, χάρτη δεμελιωδών δικαιωμάτων, την συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν αναφέρεται τίποτα για την ε, χριστιανική πλευρά της Ευρώπης. Αυτές όμως είναι οι αξίες πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε η Ευρώπη πρέπει να τις συνειδητοποιούμε και να τις ξεκαθαρίσουμε. Η δημοκρατία και το κράτος ε, δικαίου είναι εκεί ως, ε, ε, κατάσταση, όμως οι αξίες είναι αυτές. Τώρα ο Μάρκο Τσάνι για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιστεύω ότι ο τίτλος που επελέγει για αυτή τη συζήτηση έχει πετύχει 100% για να μπορέσουμε να δούμε τα προβλήματα τα οποία σήμερα αντιμετωπίζουμε. Κυρίως χρησιμοποιεί τον όρε επανείδηση, επαναθεμελίωση. Όταν ζητάτε μια επαναθεμελίωση σημαίνει ότι κάτι έχει καταστραφεί. Εδώ η Ευρώπη έχει καταστραφεί από τις πολιτικές που επιβάλλονται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρησιμοποιείται όρο όρος Ευρώπη και όχι Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ώρα να καταλάβουν οι πολίτε ότι αυτέ είναι δύο έννοιε διαφορετικέ. Η Ευρώπη είναι ένα πράγμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι άλλο. Να σταματήσουμε πια αυτή τη ρητορική, να καταστρέψουμε αυτή τη ε, ρητορική. There is no alternative. Δεν υπάρχει εναλλακτική και το μέλλον τη Ευρώπη μπορεί να είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μετά παρατίθενται τρία θεμελιώδη σημεία στα οποία πέτυχε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αξίε, διότι οι συνθήκε εδράζονται επί αξιών εντελώ εσφαλμένων ε, θα πρέπει να έχουμε δημοκρατικού θεσμού. Σήμερα το μεγαλύτερο κομμάτι των θεσμών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω δεν είναι δημοκρατική. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ένα παράδειγμα. Και να προτείνεται μια ευημερία, ευημερούσα οικονομία. Είναι σαφέ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχε όσον αφορά την οικονομική πρόοδο. Ο μοναδικό τρόπο να επαναθεμελιωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, να εγκαταλείψουμε αυτές τις συνθήκες οι οποίες χρεοκόπησαν και απέτυχαν και να επαναθεμελιωθεί σε συνεργασία Ευρώπη, ισότιμη συνεργασία μεταξύ κυρίαρχων κρατών. Αυτό είναι ο μόνος τρόπος, διότι αργά ή γρήγορα η τεράστια σύγκρουση που υπάρχει μεταξύ του κοινωνικού μοντέλου που προτείνουν συνθήκε και του κοινωνικού μοντέλου που προτείνουν οι θεσμοί, οι εθνικοί θεσμοί, θα διαφανεί. Οι συνθήκε μιλάνε για ανταγωνισμό, για αγορά, για κέρδο, για ε, διάφορα μοντέλα ε, εργασίας που είναι αντίθετα με το ε, μοντέλο των συνθηκών. Σύμφωνα με το γερμανικό μοντέλο, το Σύνταγμα τη Ιταλία, στα πρώτα άρθρα αναφέρεται στο κοινωνικό μοντέλο και μιλάει για την εργασία, προστασία τη εργασία, ένα σημαντικό στοιχείο τη παραγωγή. Αυτό σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμβαίνει. Είναι σαφέ ότι αν θέλουμε να προχωρήσουμε, ο μοναδικό τρόπο είναι να διαλύσουμε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι είναι η κορονίδα δύο εγχειρημάτων πολύ επικίνδυνων γερμανικού υπεριαλισμού και τη πειθαρχία των αγορών και συνθήκων σε εξωτερικούς δεσμούς, που είναι τυπικό των ε, ελίτ των περιφερειακών χωρών. Um, Ωραία. Τώρα ένα λεπτό Μαρία Γκραπίνη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, Επίτροπε. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ στον τίτλο, δεν έχω τίποτα εναντίον του τίτλου. Είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε επί των ουσιαστικών. Αν δεν επανεξετάσουμε, αν δεν επαναθεμελιώσουμε την Ευρώπη, θα αποτύχουμε. Πρέπει να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη που είναι ενωμένη, που βασίζεται επί αξιών. Επίτροπε, σας παρακαλώ μην παρουσιάζετε διάφορα σενάρια, μην τροφοδοτείτε τον ευρωσκεπτικισμό περαιτέρω. Εγώ έγινα πολιτικός διότι ήθελα για την χώρα μου και την Ευρωπαϊκή Ένωση όλα να βασίζονται σε αξίες. Τώρα που η χώρα μου είναι 10 χρόνια μέλος της Ένωσης, εξακολουθούμε να είμαι εκτός διάφορων χώρων. Είμαστε, είμαστε εκτός του Σέγγεν, Φερρυπίν. Οι πολίτες έχουν διάφορα καθεστώτα στα οποία πρέπει να συμμορφώνονται. Θα πρέπει να είναι ενωμένοι οι πολίτε. Θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα πάντα οι πολίτε. Ισότιμη πρόσβαση για όλου του πολίτε. Πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα στην παιδεία. Διότι ο κόσμο πρέπει να καταλάβει ότι οι πολιτικοί ηγέτε ε, εκλέγονται για να κάνουν καλέ επιλογέ για του πολίτε. Πρέπει να εκπαιδευτούν. Θα πρέπει να έχουμε αξίε που θα προωθούμε, να μα κατευθύνουν όταν αποφασίζουμε ε, ποιοι θα είναι οι ηγέτε μα. Και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι ηγέτε είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Ευχαριστούμε. Ένα λεπτό, Πέτερ Φαντάλεν. Κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο. Να σεβόμαστε αμοιβαία τις, ε, τις κουλτούρες μας. και οι εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων δεν το κάνουν αυτό. Κάποιοι μπορεί να θέλουν περισσότερη Ευρώπη και κάποιοι λιγότεροι, αλλά υποτίθεται ότι αυτοί οι λιγότεροι είναι λαϊκιστές. Δεν υπάρχει όμως βάση σε αυτή την επίκριση και αυτό έχει οδηγήσει στο Brexit. Η έλλειψη σεβασμού στην άποψη του άλλου. Πρέπει να μπορούμε να μιλάμε ο ένας τον άλλο και να σεβόμαστε την άποψη του άλλου να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα μαζί και τι όχι. Ε, και η ομάδα των φιλελευθέρων θα πρέπει να προσπαθήσει να κατανοήσει καλύτερα την γνώμη των υπολείπων. Ευχαριστώ για ένα λεπτό Πέτρο Σίλβα Περέιρα. Ευχαριστώ. Παρά τις ε, θετικές ειδήσεις του τελευταίου καιρού, ε, ας μην αυταπατώμεθα το ευρωπαϊκό όραμα ζει μια βαθιά κρίση αποτελεσμάτων με αιτίες σύγνωστες. Έχουμε ελλείμματα, ε, οργανωτικά ελλείμματα στην ημερία του ευρώ και από την άλλη μεριά έχουμε και την πολιτική λιτότητας ε, που είναι οι δύο βασικές αιτίες που υποσκάπτει τη βάση του ευρωπαϊκού project. Η κρίση αυτή όμως είναι κατά βάση μια κρίση αρχών. Με αρχή στην αρχή, στην, με, με εκείνη στην αρχή της αλληλεγγύης. Χωρίς αλληλεγγύη δεν πρόκειται να βρούμε λύση σε κανένα από τα προβλήματά μας. Οι πολίτες μας μας λένε στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις ότι θέλουν να δώσουν μια καινούργια ευκαιρία στο ευρωπαϊκό όραμα. Αλλά αυτή η ευκαιρία μπορεί να συνδεθεί μόνο με μια αλληλέγγυα κοινή λύση στα κοινά μας προβλήματα. Μια λύση που θα επιτρέψει να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα για ένα λεπτό Μίχαλ. Μίχαλ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, σε αυτή τη συζήτηση μιλήσαμε για τους πατέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιλήσαμε για τη βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι δικαιολογημένο αναφερθήκαμε και στους κανόνες της ολοκλήρωσης. Κατανοούσαν οι πατές Ευρωπαϊκής Ενώσεως ότι η δημοκρατία, η οικογένεια βασίζονται, είναι βάση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Καταλαβαίνω τι ήθελε να πει ο κύριος Βέμπερ. Δεν καταλαβαίνουμε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό χωρίς χριστιανικές αξίες και δεν μπορούμε να αποδεχθούμε να αντιμετωπίζει τη θρησκεία που έδωσε ισχύ στον ευρωπαϊκό πολιτισμό ε, να αντιμετωπίζεται με προσπάθεια φήμωσης. Πρέπει να προστατεύσουμε και την ακαιρεότητα ε, της αγοράς μας λένε. Και σήμερα ο εχθρός της ακαιρεότητας της αγοράς είναι ο προστατευτισμός των πλουσίων χωρών που εκπροσωπούνται της κυβέρνησης που κλείνουν τις αγορές εις βάρος του μέλλοντος της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ευχαριστούμε τον κύριο Τζεντόφσκι και τώρα για ένα λεπτό την Μπορτσάνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγκεκριμένε πολιτικές δυνάμεις απομακρύνονται από την Ευρώπη. Θέλουν να ερμηνεύσουν με νέο τρόπο ή να παρερμηνεύσουν την Ευρώπη, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, ε, την ισότητα που αποτελούν το υπόβαθρο της Ευρώπης. Υπάρχουν πολλές αξίες ε, στην Ευρώπη και το τελευταίο διάστημα δυστυχώς ε, ασκούνται μεγάλες πιέσεις από τις εξτρεμιστικές αντιευρωπαϊκές ε, δυνάμεις. Υπάρχουν ε, φόβοι που πολλές φορές δεν αληθεύουν, όμως τα κράτη-μέλη έχουν λόγο να, το, να φοβούνται. Ένα καλό παράδειγμα είναι η σημαία του μη φιλελευθερισμού. Υπάρχουν οι ολιγάρχες ε, αυτοί που πραγματικά κυβερνούν και εμείς ε, παρατηρούμε ακριβώς ε, πως η Ρωσία έχει όλο και περισσότερο δύναμη και επιρροή. Βλέπουμε πως λειτουργεί ο Πούτιν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να ασκήσει κάποιον έλεγχο αλλά δεν το καταφέρει. Ένα λεπτό τώρα, κυρία Πατρίτσα Τόγια. Είναι πολύ ξεκάθαρο ε, Ποιε είναι οι θεμελιώδεις αξίες αυτού του οικοδομήματος. Όσο υπάρχουν κλειδονισμοί, τόσο πιο βαθιές θα πρέπει να είναι οι ρίζες. Ε, οι αξίες όπως η δημοκρατία δεν είναι κενέ περιεχομένου, ειδικά όταν έχουμε αυταρχικές διολυστεί σε κάποια κράτη-μέλη. Ε, επίσης, όταν βλέπουμε τις συγκρούσεις στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και με σημεία σύγκρουση στο εσωτερικό, η κοινωνική δικαιοσύνη είναι ακόμα πιο αναγκαία όταν βλέπουμε τα τελευταία, ότι τα τελευταία χρόνια αυξήθηκαν οι ανισότητες και οι δυσκολίες ε, σε πολλά τμήματα του πληθυσμού. Αυτά είναι θεμέλια που εγγυώνταν ε, την ένταξη. Αυτά θα πρέπει να ενισχυθούν εν ώψη της κρίσης η Λευκή Βίβλος. Ο Γιούνκερ μας μιλάει για κάποιε υποθέσεις. Δεν νομίζω, νομίζω ότι πρέπει να επιλέξουμε τη μία ή την άλλη Ευρώπη. Ένα κράτος μέλος στην Α Ευρώπη και το άλλο, το άλλο κράτος μέλος Β, τη Β Ευρώπη. Ή θα κερδίσουμε μαζί ή θα χάσουμε χώρια. Αυτές είναι οι διανατακτικές μας. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφε Τόγια. Και τώρα α, θα επανέλθουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το λόγο έχει η κ. τη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρί χωρί μικρόφωνο. Επιτρέψτε μου κάποιες σκέψεις μόνο να σας αναφέρω σε ό,τι αφορά τη συζήτηση. Ως έφηβος ε, πήγα στην Ισπανία η οποία μόλι είχε βγει από την περίοδο τη δικτατορία και ω νεαρό από την Ολλανδία, από τι κάτω χώρε, με σοκάρισε ιδιαίτερα η κατάφορη φτώχεια στην ε, Ισπανική Ήπεθρο, όχι μόνο η φτώχεια, αν θέλετε, σε οικονομικού όρου, αλλά και η ηθική ένδυα. Η οικογενειακή βία ήταν κάτι ενδεμικό ως φαινόμενο. Τα παιδιά δεν πήγαιναν στα σχολεία, ή πήγαιναν σε άσχημα σχολεία και δεν παρακολουθούσαν καν, γιατί ήταν τα κορίτσια. Γιατί κοιτάξτε που βρίσκεται η Ισπανία σήμερα. Κοιτάξτε τι έχει πετύχει. Δεν ε, πιστεύω ότι α, αυτό το πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ισπανικός λαός το πετύχει αυτό, αλλά πιστεύω ότι στα μέτρα αυτά, χωρί να ήταν μέλη της ε, ευρωπαϊκής Ιστορία, τη Ευρωπαϊκή Ένωσης, το 1999 το 89 ο κόσμος ε, κατέρευσε, το οποίο αποτέλεσε προφανώς το πιο σημαντικό πολιτικό ε, γεγονός ε, της ζωής μου. Η Πολωνία τότε ήταν στη χειρότερη κατάσταση από την Ουκρανία. Κοιτάξτε που βρίσκεται σήμερα η Πολωνία. Νομίζω ότι η οικονομία είναι 5-6 φορές μεγαλύτερη και πιο ανθούσα από ότι η Ουκρανική. Φυσικά δεν πιστεύω ότι αυτό είναι επίτευγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο λαός της Πολωνίας το πέτυχε αυτό, αλλά είμαι βέβαιος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθησε στην επίτευξη του στόχου αυτού ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου, όχι μόνο η οικονομία, αλλά η ανεξάρτηση του δικαστικού στόματος, η ε, αξιοπιστία, η καταπολέμηση της ε, διαφθοράς. Όποιοι λένε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τίποτα παρά ερήπια, πρέπει να έχουν χάσει, να κοφεύουν τις τελευταίες, ε, τα τελευταία 30 χρόνια. Πώς έχουμε ξεχάσει αυτά τα ιστορικά επιτεύγματα. Αυτό είναι το πρώτο σημείο που υπογραμμίζω. Και αν ξέρουμε τι έχουμε να πετύχουμε μετά την κρίση αυτή, όπου η ενεργεία είναι η πιο υψηλή παραποτέ, ξέρω ότι πολλά ακόμα πρέπει να ξεπεράσουμε, αλλά τουλάχιστον ας έχουμε λίγο πιο, παρα... πιο πολύ αυτοπεποίθηση, ότι μπορούμε να πετύχουμε. Κοιτάξτε τι, ξεπέρασαν οι γονείς μας, η γενιά των παππούδων μας. Δεν μπορούμε να πτωηθούμε ψυχολογικά. Και να τονίσω και το εξής. Ε, οι αξίες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αξίες τις οποίες βασίζεται η Ένωση, κατοχυρώνοντας το άρθρο 2 της συνθήκη και οι αρχές αυτές ε, έχουν υπογραφεί, έχουν επικυρωθεί από κάθε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ναι, υπάρχουν πολιτισμικές διαφορές και υπάρχουν και κάθε είδου διαφορές, αλλά το άρθρο 2 είναι δεσμευτικό για κάθε κράτος μέλος και για κάθε φορέα στα κρατημέλη αυτά και δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί και να ξεφορτωθεί αυτή την ευθύνη πολύ απλά με επιχειρήματα πολιτισμική φύσης και νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο μιλάμε σήμερα για επανίδρυση αν θέλετε είναι επειδή έχουμε κατανοήσει ότι δεν είναι άθραυστη η Ένωση δεν ε, μπορούμε να μην να αγνοούμε τις θεμελιώδεις αξίες μας τώρα που βρίσκονται υποκριτικοί, ξέρουμε ότι θα πρέπει να αρθώσουμε το αναστημά μας και να τις προσπιστούμε πιο πολύ παραποτέ. Και θέλω να πω και ένα πράγμα σε ό,τι αφορά τις χριστιανικές αξίες της Ευρώπης. Και αυτό το λέω ως χριστιανός, ναι, ασφαλώς ο χριστιανισμός έχει τεράστιο ρόλο να διαδραματίσει και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των αξιών μας. Αλλά είμαι πάρα πολύ ε, διστακτικός ως χριστιανός να πω ότι έχουμε πνευματική ιδιοκτησία στο ευρωπαϊκό δίκαιο ως χριστιανοί. Δεν θα είμαστε εδώ χωρίς τους ομανιστές, δεν θα είμαστε εδώ που βρισκόμαστε χωρίς το διαφωτισμό. Η ίδια μου η Εκκλησία πέρασε από το διαφωτισμό, ούτε η Ράη εξέταση της Ισπανίας, ε, ξέρετε, την εφέδρα ε, άθεη. Ας αναλάβουμε λοιπόν όλες τις ευθύνες μας για αυτά που έχουμε δώσει, αλλά σεβαστούμε και την ποικιλία και την ε, πολυμορφία των αξιών μας. Δεν μπορεί κανείς να τις διεκδικήσει ούτε από κάποια πολιτική παράταξη, ούτε από κάποιο θρησκευτικό δόγμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αντιπρόεδρο και τώρα η κυρία Ντάλη από πλευρά του Συμβουλίου. Πρόεδρε, Επίτροπε, αξιότιμοι βουλευτές, σας ευχαριστώ για τα πολύτιμα σχόλιά σας που προφανώς κατέγραψα σας διαβεβαιώνω ότι ο προβληματισμός για το μέλλον της Ευρώπης θα συνεχιστεί και θα είναι πάντα ψηλά στην ατζέντα μας, από τις πρώτες προτεραιότητες. Διερευνώντας τις ε, οδούς που θα οδηγήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να λύσει τάχιστα όλα τα προβλήματα ως διαμαγείας. Και δεύτερον, θα πρέπει τα ιδεώδη μας να τα εξορροπήσουμε με κάποιες, κάποιους πρακτικούς περιορισμούς. Άρα αυτό περιορίζει τις φιλοδοξίες μας ορισμένε φορές. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές για το τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ ολοκληρώ.